κανόνες μέχρι πέρατος. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να μας βοηθήσουν να είμαστε προσεκτικοί, να μην καταργήσουμε και τα θετικά μαζί με τα αρνητικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πέρα τη συζήτηση οι ψηφοφορίες θα γίνουν σε δύο εβδομάδες από σήμερα στην Ολομέλεια των Βρυξελών. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο το πρωί στις 20 ε, Απριλίου Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 και από τις 3 το απόγευμα μέχρι τις ε, 8 ε, και μισή και από τις 9 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα πρακτικά θα δημοσιευτούν και μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο διαδίκτυο. Πέρα στις συνεδρίασεις είναι 11 η ώρα. Καλό σας βράδυ, καληνύχτα. νύχτα. <laughs>